και περνούμε σε επεξηγήσεις ψήφου. Δεν έχει ζητήσει κανείς προφορική, εάν θέλετε, γραπτός. Να αποστείλετε στην Προεδρία. Διακόπτεται η συνεδρία σήμερα τις 11.30, όπου θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.